Κυρία Κρέτσου. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι υποψήφια επίτροπος για την περιφερειακή ε, πολιτική και θέλω να ζητήσω την υποστήριξή σας. Ξέρω την διαδικασία διαπραγμάτευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές γιατί ε, καταβάλατε μια συλλογική προσπάθεια. Μετά από μια διετή διαδικασία διαπραγματεύσεων έχουμε ένα νομοθετικό ε, πακέτο. Επίσης υπάρχουν ε, νέα μέλη που έχουν μεγάλη επιτόπια πείρα και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην εργασία μας τα επόμενα έτη. Επίσης θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στον Επίτροπο Χάν, ο οποίος πραγματικά αναθεώρησε και μεταρρύθμισε αυτή την πολιτική. Η περιφερειακή πολιτική δείχνει την αλληλεγγύη μας μέσα στα πλαίσια του προτύπου κοινωνικής αγοράς και επειδή σήμερα αποζητούμε να βγούμε από την κρίση, η περιφερειακή πολιτική θα υποστηρίξει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Μας δίνει την ε, δυνατότητα να αποστείλουμε ένα μήνυμα ως προς τα ευεργετήματα της ολοκλήρωσης στο Βορρά και Νότο, στην Ανατολή και τη Δύση, τη στιγμή που ολοκληρώνουμε την ανταγωνιστική οικονομία για όλους τους πολίτες. Γι' αυτό πιστεύω ότι η περιφερειακή πολιτική θα συνεισφέρει στην ε, εργασία του κυρίου Γιούνκερ ως προς την, ε, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής μοχλεύσεων και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η πολιτική θα ορίσει και τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα της καινοτομίας, ΜΜΕ, ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ολοκλήρωση, κλιματικές αλλαγές, διευρωπαϊκά δίκτυα και ε, εξάλληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις ε, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες και αρχές σε σχέση με το τι επικρατεί είτε στις πρωτεύουσες είτε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Θα συμπεριλάβουμε και τους τοπικούς παράγοντες καθώς και τους περιφερειακούς. Μιλάμε για 270 περιφέρειες και 500, 500 εκατομμύρια πολίτες, πάνω από 500 εκατομμύρια. Χρειάζεται υποστήριξη του προϋπολογισμού. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπή από τους πλούσιους στους φτωχούς. Είμαι πεπισμένη ότι επενδύοντας την πραγματική οικονομία στους ανθρώπους, στις περιφέρειες, εάν τους βοηθήσουμε, τότε η ευρωπαϊκή οικονομία θα καταστεί πιο εύρωστη και φυσικά το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των μερών του. Ως προς τις ε, πολιτικές μου προτεραιότητες, αν διοριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να εξασφαλίσω, να βελτιστοποιήσουμε την ε, ε, συμμετοχή της περιφερειακής πολιτικής για δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Επίσης, η μεταρρύθμιση όρισε τον επενδυτικό πυλώνα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Επίσης θέλουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα για να βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, λειτουργικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα τα επόμενα 7 χρόνια και θα πρέπει ε, να ε, προωθήσουμε τις ΣΟΕΣ οι οποίες θα δώσουν θα κάνουν τη διαφορά για την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, για τους άνεργους και για τα εδάφη και τις περιφέρειες που μπορούν πιο εύκολα να αποδομηθούν. Θα ήθελα να πω ότι η ο ποιοτικός προγραμματισμός δεν θα πρέπει να διακυβευτεί. Άρα το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική πολιτική, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, έτσι ώστε οι νέες αρχές αιρεσιμότητας να τηρηθούν με βάση τις ε, ευρωπαϊκές ε, προπτικές και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Τη στιγμή που οι δημόσιοι πόροι, οι εξασθενούν, τα καλύτερα προγράμματα σημαίνουν μεγαλύτερη απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτό θα ήθελα να το κάνω σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνου ε, συναδέλφους για την τομεακή αυτή ε, πολιτική, επιζητώντας συνέργειες και υποστήριξη από κοινοτικές ε, δράσεις. Θα ήθελα να με υποστηρίξετε Επίσης, αποστέλλοντας ένα μήνυμα στα κράτη-μέλη, η περίοδος προγραμματισμού 14-20 δεν αφορά ένα πρότυπο business as usual. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι... Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και όσον αφορά τις υποχρεώσεις νομίζω ότι οι βασικοί δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που λαμβάνουν. Πρόκειται για τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Θα πρέπει να δείξουμε τη δέσμευσή μας στο ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό με αυτά αποτελέσματα. Μαζί είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Όπως προβλέπετε από τον κανονισμό θα υποβάλλω στην Ρέτζη του χρόνου την έκθεση της έκβασης των διαπραγματεύσεων, αν διοριστώ ως προς την βέλτιστη διακυβέρνηση και την ε, θεσμική δυναμική και ικανότητα, πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό από τα χρήματα και απαράβατος όρος για να επιτύχουμε. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή διοίκηση διοικητικά μέσα, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει υποστήριξη για τη θεσμική ικανότητα στα νέα, με τα νέα προγράμματα και να υποστηρίξουμε τα κράτη κατά την επόμενη περίοδο. Χρειάζονται εταιρικές σχέσεις και συνέργεια δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Επίσης χρειάζονται εταιρικέ σχέσεις υψηλής ποιότητας για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Πολλά μπορούμε να μάθουμε από τις βέλτιστες πρακτικές των περιφερειών, των πόλεων, των τοπικών αρχών και των ΜΚΙΟ θα κάνω πλήρη χρήση των νέων δυνατοτήτων από το, τα αστικά δίκτυα μέσα στα πλαίσια της ανταλλαγής ε, εμπειριών. Επίσης, ε, δεν απλουστεύουμε πάντα τις πολιτικές μας υπέρ των δικαιούχων και γι' αυτό θα πρέπει να ε, εισακουστούν οι ΜΜΕ μέσω της υποστήριξης με αυτή την ε, πολιτική, γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Το ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει δυνατότητες να υποστηρίξουμε τους δικαιούχους και θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τηρηθούν αυτές οι αρχές. Επειδή η πολιτική συνοχής αποτελεί το 1 τρίτον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα προσδώσω μεγάλη σημασία στα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει καλή διαχείριση των διαρθρωτικών ε, ταμείων με βάση την ε, χρηστή οικονομική διαχείριση. Θα υπάρχει μηδενική ανοχή στην απάτη. Γι' αυτό θα ήθελα να δούμε καλύτερα την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής. Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Επίτροπή σας για να δω πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα ζητήματα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και με τους πολίτες, διότι νομίζω ότι δεν μπορούμε πάντα να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Ως προς την αποδοτικότητα της πολιτικής θα ληφθεί υπόψη στο επόμενο ε, νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2020 θα ήθελα να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από τα πρωταρχικά στάδια, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στις πολιτικές κατευθυντηρίες γραμμές. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ε, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Άρα θα ήθελα να επιδοθούμε σε έναν επικοδομητικό πολιτικό διάλογο με βάση τα, το χαρτοφυλάκιό μου για την χρηστή διακυβέρνηση. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου θα πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και κοινού στόχους για να συνεργαστούμε προς συμφέρον των πολιτών. Γι' αυτό θα συνεργαστώ με σας έτσι ώστε να φτάσουμε στους κοινού στόχου. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για μια κοινή συζήτηση και μια κοινή προσπάθεια να είναι αποτελεσματική η πολιτική αυτή.